Τώρα θα συζητήσουμε έξι σχέδια ψηφίσματος για την Συρία, ιδίω δε την υπόθεση του Μονάδ Αρχασανή. Θα δώσω το λόγο στους συντάκτες. Η κυρία Φρανσίσκα Μπράτζινερ, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Θέλω να μιλήσω για τον κύριο Μουχάμεντ Αρχασάνη, ο οποίος φυλακίστηκε γιατί υποστήριξε τα δικαιώματα του ανθρώπου των συμπατριωτών του στη Συρία έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί παρατήρησε όλες τις δίκες ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ασφαλεία και έκανε τακτικές αξιολογήσεις των συνθήκων κράτηση στη Συρία. Ο ίδιο τώρα είναι κρατούμενος και στη φυλακή. Ζητήσαμε από τη Συρία να τηρήσει τις υποχρεώσει της και να σεβαστεί το Διεθνές Σύμφωνο Πολιτικών και Αστικών Δικαιωμάτων και τη σύμβαση τη σύμβαση της Γενέβης κατά, τη, κατά της Δημοκρατίας. Συμβάσεις των οποίων είναι κατά ε, των βασανιστήριων, συμβάσεις κατά τις οποίες είναι μέλος και να απελευθερώσει τους κρατούμενους Δύση, τους αγωνιστές για τα δικαιώματα του ανθρώπου που βρίσκονται στη φυλακή. Επίσης ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης να προτείνει την υιοθέτηση ενός οδικού χάρτη πριν ολοκληρωθεί η Συμφωνία Σύνδεσης που θα παρέχει στόχους για τη βελτίωση του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούμε επίσης από τη Συρία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και θεωρούμε ότι αυτό είναι και δική μας ευθύνη, ευθύνη της Ένωσης ιδιαίτερα να εξασφαλίσει ότι η Συμφωνία Σύνδεσης θα επιτρέψει την εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας για το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Βαρονίκ Κέιζερ. Για πόσο χρόνο, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι ε, είμαι αρκετά μπερδεμένη και θλιμμένη και απογοητευμένη. Γιατί μπερδεμένη, γιατί αναμφισβήτητα στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων η Συρία τα τελευταία δύο χρόνια ε, έκανε μεγάλα βήματα πρόοδου, μπήκε στην Ένωση για τη Μεσόγειο, πολλές φορές χρησιμεύει σαν διαμεσολαβητή σε δύσκολες διεθνείς συνθήκες όπως πολύ πρόσφατα κατά τη σύλληψη μιας νεαρής στο Ιράν και μπορώ να πω ότι το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία σύνδεσης που δεν έχει υπογραφεί ακόμα αλλά που μπορεί να υπογραφεί σύντομα το γεγονό ότι ξεκίνησε ξανά αυτή η διαδικασία είναι από μόνο του κάτι πολύ θετικό. Τώρα στο εσωτερικό επίπεδο είναι γεγονό ότι και εδώ έχουμε πολύ καλά ε, σημάδια από τη Συρία. Ε, ασχολούνται με πρόσφυγε από το Ιράκ, έχουν αναλάβει σημαντικέ δεσμεύσει, απελευθέρωσαν Κούρδους. Αλλά στο επίπεδο των πολιτικών ελευθεριών και του πλουραλισμού δεν έχουμε ε, κάτι να, να πούμε θετικό. Και πραγματικά εκφράζω τη λυπή μου για την επανειλημμένη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την φυλάκιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλές φορές τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να ε, παρεύουμε για την ε, απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Ε, μερικές φορές το καταφέραμε να απελευθερωθούν, αλλά απομένουν ακόμα στι Συριακέ φυλακέ άνθρωποι όπως ο Λαμπονί, ο Αλμπουινί και τώρα ο... Ε, Αλ Χασανή. Πραγματικά θέλουμε να βγάλουμε τη Συρία από την ε, απομόνωση που είχε βρεθεί ε, στο παρελθόν. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για την διεθνή σκηνή, αλλά και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά έλεος πια για την ίδια την εικόνα της. Ε, θα πρέπει πλέον η Συρία να δεχτεί ε, τον πολιτικό πλουραλισμό και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων και επιτέλους έλεος ας απελευθερώσει τους πολιτικούς ε, κρατούμενους, ας σεβαστεί την συνθήκη για τα βασανιστήρια. Είναι προς το συμφέρον της Συρίας και προς το συμφέρον της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ασία Ανατολή πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Βέμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έχουμε πάλι έναν αγωνιστή τον οποίο θέρετα ε, κρατούν οι αρχές της Συρίας. Και η μόνη του επιθυμία ήταν να προστατεύει τους ανθρώπους για να μπορούν να εκφράζουν εύκολα και άνετα τις απόψεις τους ε, το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη. Για πάνω από πέντε χρόνια του είχαν απαγορεύσει να ταξιδεύει. Είχε το γραφείο του εκεί οι τηλεπικοινωνίες και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ήταν μόνιμα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις ασφαλείας. Μετά από πολλές εβδομάδες όπου τον παρενοχλούσαν τελικά συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας και κατόπιν καταδικάστηκε για διάφορα ποινικά αδικήματα που όλα έχουν σχέση με το δικαίωμά του της ελεύθερης έκφρασης απόψεων. Και όταν μιλάμε για αυθαίρετη κράτηση, ας μην ξεχνάμε τον κύριο Αλαμπανή, ο οποίος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για εκείνα τα οποία τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι είναι η ειρηνική έκφραση των πολιτικών του απόψεων. Η κυβέρνηση της ε, ε, Συρίας πρέπει να απελευθερώσει αυτούς τους δύο αλλά και όλους τους άλλους πολιτικούς κρατουμένους αμελητή και χωρίς ε, προϋποθέσεις και ε, φυλάσσοντας ε, την ψυχική τους ε, και την σωματική τους ακαιρεότητα. Οι αρχές της Συρίας πρέπει να καταργήσουν όλες τις μορφές παρενόχλησης απέναντι σε όλους τους αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και αυτό σε συμφωνία με τη δήλωση περί υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Τάνοκ. Βέβαια, η Συρία παίζει βασικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και ε, στις προσπάθειες να ε, μειωθεί η ένταση με το ε, Ιράν. Ταυτόχρονα η Συρία ε, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το Λίβανο. Είναι ένα καθεστώς κοσμικό βεβαίως και παραμένει το μόνο σημείο, το μόνο ισχυρό σημείο του παλιού ισχυρού Μπάθ προστατεύονται κατά κάποιο τρόπο τα δικαιώματα των γυναικών, για παράδειγμα. Παραμένει, ωστόσο, ε, μία μονοκομματική δικτατορία. Ο Αλ Χασανή είναι ένας αγωνιστής για τα δικαιώματα των ανθρώπου που αδίκως φυλακίζεται. Αν θέλει να πιστέψουμε ότι η Συρία αλλάζει, η χώρα αυτή πρέπει να απελευθερώσει άμεσα τον κύριο Αλ Χασανή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόλχολα, δύο λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τίθεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή διότι ε, πρόκειται να υπογραφεί συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συρία και ως εκ τούτου θεωρώ ότι η Συρία πρέπει να μπορεί να επιδείξει ουσιαστική βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη χώρα αυτή. Γιατί όσα έγιναν μέχρι τώρα δεν αρκούν. Ο ε, νομικός ε, κύριος Χασάνη συνελήφθη και αυτό με βάση ψευδομαρτυρίες. Πέρυσι και πρόπερσι εμείς ταχθήκαμε υπέρ των αγωνιστών ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, αλλά αυτοί εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή. Η Συρία ε, πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα όσον αφορά ε, την ασφάλεια στη χώρα αυτή. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι το βρίσκω ιδιαίτερα λυπηρό το να μην σεβόμαστε και να μην εφαρμόζουμε στην περίπτωση της Συρίας τα κριτήρια της ελευθερίας διότι για να υπάρξει συμφωνία σύνδεσης ε, πρέπει να διαπιστωθεί ότι διαφυλάσσονται πράγματι τα κριτήρια της ελευθερίας. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο δεν ε, είναι μία απομονωμένη νησίδα, όλα είναι αλληλένδετα και δεν πρέπει να αγνοούμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο αν κρατάμε τα μάτια ανοιχτά ε, θα μπορούμε να καταστήσουμε τη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο ανεκτή. Ευχαριστώ, πολύ. Για ένα μισή λεπτό. Ε, η κυρία ε, ο Ευχαριστώ πολύ. Ο Μοχάμεντ Αλ Χασάνι. Ένας από μια από τις ηγετικές προσωπικότητες για στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, τον Ιούλιο συνελήφθη, δικάστηκε και κλεισμένο των θυρών, κατηγορήθηκε για υπονόμευση ε, του εθνικού ε, κύρους για υπόσκεψη εθνικού αισθήματο και διασπορά ψευδών ειδήσεων. δεν του δόθηκε η άδεια να φύγει από τη χώρα. Ε, παρακολουθούνταν συνεχώς οι δραστηριότητες τους του για, την, για τον έλεγχο του ε, Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου στην ασφαλεία και ασφαλείας και πραγματικά είναι πάρα πολύ ενσυχετικό ότι δεν υπάρχει καθόλου πρόοδος ε, όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, η Συρία πρέπει να σεβαστεί τη Σύμβαση των ΕΕ για την απαγόρευση των βασανιστήριων και γενικά την κακομεταχείριση των κρατουμένων. Ε, αν λάβει κανεί υπόψη του δεσμού που υπάρχουν ανάμεσα στη χώρα αυτή και την Ευρώπη και το σημαντικότερο ρόλο που έχει η Συρία για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ε, βάσει όλων αυτών, είμαι πεπισμένη ότι η Συρία μπορεί να προοδεύσει στον τομέα αυτό και έτσι να προοδεύσει η δημοκρατία σε ολόκληρη την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Ομπερμάιερ. Ε, αυτή την πρόταση ψηφίσματος την βρίσκω σωστή. Ε, πρόκειται να υπάρξει σύνδεση και ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να ε, προστατεύσουμε τις οικογένειες του κατηγορουμένου, του αγωνιστή Αλχασάνη και το άρθρο 2. Και εξάλλου αυτό πρέπει να το πράξουμε γιατί εμεί, ως Ευρωπαίοι που είχαμε μια οδυνηρή ε, ιστορία ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδώ και δύο δεκαετίε μόνο κατέρευσαν αυτά τα κομμουνιστικά συστήματα. Εδώ όμως θέλω να σας προειδοποιήσω και για το εξή. Να μην κλείνουμε τα μάτια όταν στη γειτονιά της Συρίας, στην Τουρκία συγκεκριμένα, αγνοούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μάλλον ε, που η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα όπου η νομολογία, η προστασία των μενοτήτων, η άνεξη θρησκεία όλα αυτά είναι ελληματικά ακόμα και εάν υπάρχει μια εξοραϊσμένη συγκεκριμένη έκθεση, η περίφημη έκθεση Αχτισάρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ολοκληρώνονται έτσι οι αγορητές. Ο κύριος Πόσελτ όμως έχει ξαναζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολύ επικριτικό πνεύμα την κατάσταση στην Τουρκία. Είναι δικτατορία και αστυνομικό καθεστώ και πρέπει να απελευθερωθεί ο κύριο Αλχασάνη. Πρέπει όμω ε, να κατανοήσουμε ότι ο πρόεδρο Ασάντ, ο οποίο ανοίγεται τώρα και ο πατέρα του, παραδείγματο χάρη, ε, την συμβίωση μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών την καλλιέργησαν και ο ε, Νταού, το επίσκοπος Νταού, γνωστός ε, χριστιανός στη Συρία, είπε ότι οι χριστιανοί στη Συρία αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς από ότι στο Ιράκ που υποτίθεται στηρίζουν οι δυτικέ δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν διαφοροποιημένη πρέπει να είναι η στάση μας στη Συρία. Εντάξει, να στυλιτεύουμε την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως να στηρίζουμε τη χώρα σε αυτό το άνοιγμα που κάνει. Ε, και σαφώς να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιες θετικές τάσεις τις οποίες πρέπει να στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ξαναδώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή συμμερίζεται τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δικαιωμάτων των ανθρώπων στη Συρία. Η εκτίμησή μα είναι ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε του τελευταίου μήνε. Υπάρχουν περισσότερε αυθαίρετε ε, συλλήψει, παραβίαση των δικαιωμάτων των αγωνιστών. Ο κ. Μοχάμετ Αλ Χασάνη στι 30 Αυγούστου συνελήφθη. Πρόκειται για έναν γνωστό δικηγόρο οργανώσεων δικαιωμάτων ανθρώπων στη Συρία και μέλο του δικηγορικού συλλόγου τη Δαμασκού για 15 χρόνια. Ο κ. Χασάνη είναι Αγωνιστή των Ευρωπαίων δικαιωμάτων και φαντάζεται κανεί ότι η σύλληψή του είχε πολιτική, πολιτικά αίτια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη εξέφρασε τι ανησυχίες τη προ τι αρχέ Συρία. Η Συρία πρέπει να τηρήσει τι διεθνεί δεσμεύσει τη, ιδίως την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων και το Διεθνέ Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, των οποίων μέλο συμβαλόμενο είναι η Συρία. Η Επιτροπή ε, ζήτησε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής στη Ρωμασκοκή, οι πρεσβείες των κρατών μελών συζητούν την ε, δυνατότητα να λειτουργήσουν, να ζητήσουν από αγωνιστές των δικαιών δικαιωμάτων να υποστηριχθούν δικηγορικά από εμά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει τήρηση, των, ε, σεβασμός ε, από των βασικών αρχών της δικαιοσύνη από ότι τα δικαστήρια που θα τους κρίνουν. Πρέπει να ζητήσουμε από τα ευρωπαϊκά εργαλεία από τη υποστήριξη, να δώσουμε υποστήριξη στις οικογένειες και τα άτομα από τον προπολογισμό της Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και πιστεύουμε ότι η Ένωση θα έχει ε, μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβαση στη Συρία αν είχε υπογραφεί η Συμφωνία Σύνδεσης. Χαίρο διότι η Προεδρία εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογραφεί η συμφωνία αυτή τι επόμενε εβδομάδε. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει τη δημιουργία ενό μόνιμου διαλόγου για να προωθήσουμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.